welcome. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στην πρώτη συνεδρίαση τη Επιτροπής Οικονομικών της ε, θητεία αυτής, μετά βεβαίω την σύστασή μα σε σώμα. Λοιπόν, έγκριση ημερήσια διάταξη αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. ευχαριστώ. Μετά έχω μια ανακοίνωσούλα για τα γλωσσικά. Όπως ξέρετε, ο κώδικας περί πολυγλωσσίας αφορά τη μετάφραση και τη διερμηνία στο Κοινοβούλιο. Μία απέτηση είναι ότι η Επιτροπή μας, όπως και όλες οι Επιτροπές, θα πρέπει να τηρεί ένα προφίλ γλωσσών με βάση τις ανάγκες των μελών. Η διαχείριση του είναι ευθύνη της γραμματείας. Για τον σκοπό αυτό έχουν προωθηθεί στην διοίκηση προφίλ με 12, 16, 20 και 23 γλώσσες όταν λοιπόν έχουμε συνεδριάσεις, ε, οι αίθουσες κατά κανόνα ανταποκρίνονται στον αριθμό των καμπίνων διερμηνίας. Διαβεβαιώ τα μέλη ότι η Επιτροπή μας είναι μία από τις μεγάλες επιτροπές και έχει κατά κανόνα υπηρεσίες διερμηνίας, όμως ε, μερικές φορές ε, θα είναι αναπόφευκτο να έχουμε μειωμένε γλώσσε, παραδείγματο χάρη για έκτακτε συνεδριάσει σε Στρασβούργο και Βρυξέλλε. Οπότε η Γραμματεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα γλωσσικά προφίλ και να τα προσαρμόζει όταν αυτό είναι αναγκαίο. Αλλά σήμερα νομίζω έχουμε πλήρε καθιστώ, έτσι. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε περνάμε τώρα στο σημείο 3. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Κένιγκ, πρόεδρο του ενιαίου μηχανισμού ε, διάσωσης στην πρώτη ακρόαση για αυτήν την θητεία με βάση τον κανονισμό που συνέστησε το Συστημικό Συμβούλιο Σταθερότητας ε, και για να υπάρχει δημοκρατική λόγοδοσία. Η κυρία Κένεγκη είχε έρθει τελευταία φορά στις 2 Απριλίου στην Επιτροπή μας. Σήμερα παρουσιάζει την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου της για το 2018 με στόχο τα σχέδια διασώσεων τράπεζων, το υφιστάμενο πλαίσιο, μέτρα διαχείρισης κρίσης και το ενιαίο ταμείο διάσωσης. Βεβαίως είμαι σίγουρος ότι οι βουλευτές ε, επί τη ευκαιρία θα αναφερθούν και σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα, γενικότερα την Τραπεζική Ένωση και τις αρμοδιότητες ε, του Συμβουλίου αυτού, οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή ανταλλαγή απόψεων. Κυρία Κένικ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Με κολακεύετε που στην πρώτη σας συνεδρίαση με καλέσατε ε, έλεγα ότι είναι η έλεγα και περίμενα την τελευταία εβδομάδα πριν πάμε για διακοπές πρώτα απ' όλα ε, να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για την επανεκλογή σας Αναμένω την συνεργασία μαζί σας ε, στην θητεία αυτή γιατί βεβαίως η λογοδοσία, η διαφάνεια είναι κάτι που παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και για εμένα είστε και πρέσβης ε, μιας δουλειάς η οποία είναι αρκετά μοναδική και πρέπει να την εξηγείτε στους ψηφοφόρους σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια γενική εικόνα του τι κάνουμε, θα είμαι πολύ σύντομη, μετά να κάνω μια σύνοψη των τομέων στους οποίους έχει σημειωθεί πρόοδος, να σας πω πού βρισκόμαστε και τέλος, επί τη ευκαιρία, θα εξετάσουμε λίγο το μέλλον ε, σε ζητήματα που θεωρώ ότι είναι βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις για εμάς αλλά και γενικότερα και για εσάς, ε, για το Συμβούλιο στην θητεία αυτή και οπωσδήποτε θα σας παραπέμψω στην ετήσια έκθεσή μας ε, την οποία είμαι σίγουρη ότι την έχετε διαβάσει και την ξέρετε απ' έξω. Πρώτα απ' όλα για εμάς. Νομίζω ότι η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης ε, ήταν νομίζω θεμέλιος λίθος της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράχ του 2008. Η Τραπεζική Ένωση σχεδιάστηκε με τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι ο ενιαίος υποπτικός μηχανισμός Φραγκφούρτη, ο άλλος πυλώνας ο ενιαίος μηχανισμός ε, διάσωσης ε, με το Συμβουλίο μας και ο τρίτος ακόμα είναι η υποκατασκευή ε, ήταν ένα σχέδιο κοινών εγγυήσεων των καταθέσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το Συμβουλίο μας βασίζεται και αυτό είναι ήδη κάτι στο οποίο θα πρέπει να εργαστούμε. Βασίζεται στους κανονισμούς BRRD και SRMA, τους δύο αυτούς κανονισμούς και καθώς αρχίζαμε να τους εφαρμόζουμε Ταυτόχρονα εσείς το Συμβούλιο ή η Κομισιόν ήδη εργάζεστε σε ένα νέο τραπεζικό πακέτο το οποίο ετέθη ενισχύ ε, στα τέλη του περασμένου έτους και το οποίο πρέπει τώρα να εφαρμόσουμε. Θα επανέλθω λοιπόν στη δουλειά μας σε λίγο, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κάτι ε, το οποίο ε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι παρεξηγημένο το σκεπτικό της διάσωσης είναι, για να το πω απλά, να διασφαλίσουμε ότι μια τράπεζα η οποία θα έχει προβλήματα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί με τρόπο αποτελεσματικό με τον χαμηλότερο δυνατό αντίκτυπο στον φορολογούμενο, δηλαδή όχι άλλες διασώσεις και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την ζημία στην ευρύτερη οικονομία. Οι περισσότερες τράπεζες και έχουμε γύρω στις 3.000 από αυτές, κατά κανόνα εμπίπτουν στις εθνικές διατάξεις περί χρεοκοπίας. Είναι μικρές, δεν έχουν κρίσιμη σημασία και δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οπότε εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις περί χρεοκοπίας όπως οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Όμως για τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες η χρεοκοπία των οποίων θα επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία, έχουμε αυτήν την νέα έννοια της διάσωσης, η οποία είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας και δεν είναι, είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι κάποιο είδους πανάκια που μπορεί να άρει όλε οι συνέπειε μια τράπεζα η οποία χρεοκοπεί. Γιατί βεβαίως σε αυτήν την περίπτωση έχουμε ζημίες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν επί της αρχής από μετόχους και ομολογιούχους και όχι από το γενικό κοινό. Αυτά κάνουμε σε γενικές γραμμές ε, και για να είμαι και δίκαιοι στην περίπτωση της Banco Popular πριν από δύο χρόνια δείξαμε το πλαίσιο αυτό επί της αρχής λειτουργεί. Αντιμετωπίσαμε επιτυχώς το 2017 την πρώτη αυτή περίπτωση, προστατεύσαμε τον Ισπανό φορολογούμενο, διασφαλίσαμε την σταθερότητα του στήματος πέρσι το καλοκαίρι και ε, πριν με ρωτήσετε αν έχει οριστικοποιηθεί σας απαντώ όχι γιατί βεβαίως μετά από αυτό μετά από την εξέταση του εάν η διάσωση αυτή ήταν ε, δίκαια δηλαδή εάν επρόκειτο περί ε, ως προς αυτό ε, ακόμα γίνονται οι δημόσιες ακροάσεις. Αναλύουμε τα σχετικά σχόλια και ελπίζουμε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο τελευταίο αυτό σκέλος μέχρι το τέλος του έτους. Το αργότερο αρχές του επομένου έτους. Εντάξει, το συντομότερο δυνατόν, αλλά πάντα με ποιότητα. Και δεύτερον, για να τελειώσουμε με το θέμα της Banco Popular, καταφέραμε να οικοδομήσουμε το ταμείο αυτό διάσωσης, ε, το οποίο χρηματοδοτεί ο κλάδος. Έχουμε ένα ταμείο το οποίο υπάρχει εδώ και τέσσερα χρόνια. Έχουμε γύρω στα 33 δισεκατομμύρια και θα πετύχουμε τον στόχο του 1% των καταθέσεων μέχρι το 2023 που θα είναι δηλαδή γύρω στα 60 δισεκατομμύρια ίσως και λίγο παραπάνω. Τέλος. Έχουμε αναπτύξει σχέδια για όλους τους τραπεζικούς ομίλους ε, της αρμοδιότητός μας και συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τα σχέδια αυτά έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν να διασωθούν. Και για κάποιους, ε, αν θέλετε να κάνετε τα μαθηματικά, έχουμε 109 σχέδια για τραπεζικούς ομίλους Έχουμε 127 τράπεζες ή ομίλους, αν θέλετε, αρμοδιότητός μας, αλλά 111 σε κάποιες περιπτώσεις μετράνε δύο φορές. Δηλαδή μια τράπεζα είναι κατ' ουσίαν θυγατρική μιας άλλης, οπότε είναι 111 οι όμιλοι. Οπότε τώρα το γενικό πλαίσιο υπάρχει περνάμε από την ανάπτυξη της πολιτικής στην εφαρμογή και στη δράση. Έχουμε συνεργαστεί με τον κλάδο και τις εθνικές αρχές και έτσι διαμορφώνονται αυτές οι πολιτικές, να πτήσουμε έγγραφα κατευθύνσεων, ένα επιχειρησιακό πλαίσιο και τέλος, και αυτό βλέπετε και στην έκθεση, οι τράπεζες θα πρέπει να φροντίσουν. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι αν θέλετε αναπτύσσουμε τις απαιτήσει, τις προθεσμίες και μόνο εάν κάτι τέτοιο δεν είναι επιτυχές περνάμε σε μια διαδικασία παράβαση. Δεν λέμε εμείς ε, τι μορφή θα πρέπει να έχει η τράπεζα. Το ο κανονισμός ε, είναι πιθανώς ε, το πιο γνωστό νομοθέτημα. Λέμε ότι θα πρέπει οι τράπεζες να έχουν επαρκή κεφάλαια για να απορροφήσουν τις ζημιές και να ανακεφαλαιοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτές οι μόνες απαιτήσεις. Κλείνουμε το κενό βήμα-βήμα, αλλά έχουμε ακόμα μία μεταβατική περίοδο που χρειάζεται. Άλλα εμπόδια, για να τα αναφέρω έτσι επιτροχάδιν, οι δομές των ομίλων, είναι μάλλον ένα θέμα το οποίο συζητάμε συνεχώς. Κάποιοι όμιλοι είναι τόσο υπερίπλοκοι και έχουν τόσες μονάδες που πρέπει ακριβώς να δούμε πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα. Αποτελεσματικά συνδεδεμένα συστήματα πληροφορικής, κατά το οποίο πρέπει να γίνεται διαρκώς, πρέπει να γίνει περισσότερο επιχειρησιακή συνέχεια. Εδώ πέρα έχουν γίνει πολλά τουλάχιστον ε, στο να υπάρχει η απαιτούμενη βάση για κάτι τέτοιο, οπότε πράγματι σημειώνεται πρόοδος ως μια αφετηρία για την απαιτούμενη διαφάνεια και βεβαίως ε, διακυβέρνηση, επικοινωνία κτλ. Θα μπορούσα να συνεχίσω και είμαι σίγουρη ότι θα ρωτήσετε. Έχουμε εργαστεί και θα συνεργαστούμε και θα εργαστούμε και στο μέλλον έτσι ώστε ο κάθε όμιλος να έχει κάποια προγράμματα και απαιτήσει. Ε, το κάνουμε αυτό το 18, το 19 και θα το κάνουμε και στο μέλλον. ταυτόχρονα ε, εξεργαζόμαστε ένα έγγραφο που θα ανέβει στην σελίδα μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, να βιαστώ. Το οποίο αναφέρει τις δικές μας προσδοκίες από τις τράπεζες, οπότε υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση για όλες τι τράπεζε. Τι σημαίνει δηλαδή να είναι σε, η τράπεζα σε θέση να ανταποκριθεί. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Αυτά θα έλεγα ότι είναι η καθημερινή μα δουλειά. Αλλά πρέπει να βελτιώσουμε και το πλαίσιο για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, ένα θέμα είναι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών από κάτι που είναι ιδέα να περάσει στην πραγματικότητα και οι τράπεζες επίσης πρέπει να περάσουν στο Έμπρελ σε μια ευρωπαϊκή ε, κεφαλαία αγορά και να μην χρειάζεται να καταφεύγουν σε εμάς ή αλλού. Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσουμε το πακέτο μείωσης του κινδύνου. Κάποια μέτρα του πακέτου αυτού οπωσδήποτε για το μέλλον είναι η καλύτερη ποιότητα, ποσότητα των κεφαλαίων αυτών, αλλά είναι ένα περίπλοκο θέμα και οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη και αν μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται βήμα-βήμα. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να γίνει πραγματικότητα για να μειωθεί ή η η απόκληση των εθνικών νόμων περί χρεοκοπίας. Είναι σημαντικό αυτό τουλάχιστον να υπάρχει μια ε, εναρμονισμένη διοικητική διαδικασία για τις τράπεζες οι οποίες πηγαίνουν προς χρεοκοπία. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ε, σκεφτούμε έτσι ευρύτερα. Θα μπορούσαμε οπωσδήποτε να δούμε στενότερα το αμερικανικό μοντέλο, το FDIC, και να καταλήξουμε με κάτι ανάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω αυτό θα ήταν ένα λογικό επόμενο βήμα και τέλος, ε, κάτω που δεν αφορά τόσο πολύ εσάς, αλλά όλους εμάς, η ρευστότητα στην διάσωση είναι στο μέσο που έχουμε αναφέρει, είναι ένα βασικό κενό στο πλαίσιό μας και εδώ υπάρχει ακόμα έλλειψη σε μια ουσιαστική απάντηση. Εγώ θα επαναλάβω το παλαιό μου επιχείρημα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με εναρμονισμένη δράση μεταξύ κρατών μελών και κεντρικών τραπεζών που είναι αυτοί οι οποίοι παρέχουν στην τελική ανάγκη ρευστότητα. Και για να αναφερθώ, οι ε, κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ στην προηγούμενη θητεία δεν πρέπει να ξεχαστούν και ε, οπότε θα σταματήσω και θα περιμένω τις ερωτήσεις σας ευχαριστώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας πολύ ενδιαφέρουσα Έχουμε τα χρήματα, πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Και ρευστοποίηση να λαμβάνει η χώρα με τον σωστό τρόπο. Γιατί είναι κάτι που έχει κόστος. Η εξυγίανση έχει κόστος. Και έχουμε κενά εκεί. Στο πλαίσιό μας και είναι σημαντικό με αυτή την ευκαιρία και το διάλογο να το σκεφτούμε. Ας ακούσουμε ομιλητές. Μάρκος Φέρμπερ για το ΕΛΚ. Πέντε λεπτά για ερωτήσεις και μετά απαντήσεις. Και μετά δεύτερο γύρο, αν επιτρέψει ο χρόνος. Ο Μάρκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Κένικ, χαίρομαι που ξαναήρθατε και σας καλωσορίζω εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στο νέο Κοινοβούλιο. Ε, ε, χαίρομαι για τη συνεργασία μαζί σας. Βεβαίως χαιρόμαστε όταν δεν έχετε καμία δουλειά να κάνετε, γιατί σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει καμία τράπεζα. Αλλά κάποιος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου πριν από 1,5 χρόνο για το όργανο το οποίο διοικείται, το οποίο ανέφερε διάφορα σημεία κριτικής. Το ένα αφορά την υποστελέχωση, αλλά και την ελληπή μετάδοση δεδομένων μεταξύ επιχειρηματικών τραπεζών, εθνικών εποπτικών αρχών και του SRB. Και αυτό οδηγεί στο ότι ε, εσείς... Ε, σε σημαντικούς τομείς τη εργασίας σας που αφορούν την ανάλυση, την αξιοπιστία και την ε, δυνατότητα διάσωσης ε, τραπεζών υπάρχουν πράγματα οποία ακόμη παραμένουν ζητούμενα. Δηλαδή δεν υπάρχουν για όλες τις τράπεζες πλήρη σχέδια διάσωσης, ανάλυση των σχετικών παραγόντων. Αυτά όμως είναι η βασική σας δουλειά. Έχει περάσει 1,5 χρόνος. Τι μπορείτε να μας πείτε λοιπόν για αυτά, τι έχει γίνει έκτοτε. Κοιτάξτε, το τέλος του 2016 απεφάνθη το ελεκτικό συνέδριο. Είμαστε σε εμβριακή φάση. Έκτοτε προσλάβαμε σχεδόν το διπλάσιο προσωπικό. 400 είναι ο στόχος μας. Τώρα είμαστε 345. Και τώρα έχουμε νέο κατάλογο για προσλήψεις και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε 400 στο τέλος του έτους. Είναι θέμα το προσωπικό. Για τα στοιχεία έχουμε τεράστια βελτίωση όσον αφορά τα δεδομένα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τις Εθνικές Αρχές. Πάντα έχουμε κάποιες επιθυμίες για βελτίωση, όμως είναι άριστη η συνεργασία τα πλήρη σχέδια εξυγένσης. Πάντα έχουμε ένα ευχολόγιο για τα επόμενα βήματα. Και όταν απεφάνθη το ρεκτικό συνέδριο δεν είχαμε πλήρη σχέδια εξυγένσης. Είχαμε έναν πρώτο γύρο σχεδίων. Έκτοτε έχουμε μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε συγκεκριμένες συζητήσεις για τη δυνατότητα εξυγίανσης Ακούγονται ιδέες όμως στη συζήτηση που χρειάζουν σταδιακή επεξεργασία. Κάναμε αρκετά. Όχι στο βαθμό που θα ήθελα, αλλά ε, δύο χρόνια μετά επιστρέφει το ελεκτικό συνέδριο και θα έχουμε νέα έκθεση να αφορά τι επιδόσει και ελπίζω ότι εκεί θα διαπιστωθούν οι βελτιώσεις. Ποτέ δεν πίστευα ότι έχουμε τόσο συχνά αυτέ τι ε, εκθέσει του ελεκτικού συνεδρίου. Έχω ακόμα χρόνο κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω το ερώτημα το οποίο με ενδιαφέρει το αναφέρατε κάπως γενικώ. Υπάρχουν τώρα για όλα τα πιστοτικά ιδρύματα σχετικά σχέδια εξυγένσης ή υπάρχουν λήψεις. Κοιτάξτε, έχουμε δύο-τρει υποθέσει που χρειάζονται βαθιά αναδιάθρωση και εκεί έχουμε αναβάλει την απόφαση. Αλλά για όλου του μήλους υπάρχουν σχέδια. Μπορεί να υπάρξει διάσωση ε, για όλους. Όχι, έχουν κάποιες ε, απαιτήσει, χρειάζεται κάποια δουλειά, πρέπει να εφαρμόσουν κάποια μέτρα, να επεξεργαστούν τα έμεραλ κλπ. Αλλά όλα προχωρούν. Ευχαριστώ. Φερνάντες για τους σοσιαλιστές. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια, η οποία ελπίζω να συνεχίσει να είναι καρποφόρα για τα επόμενα χρόνια. Δύο ερωτήσεις. Δεν θα επιμείνω ως προς την ανάγκη να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Άνωση. Το είπατε εσείς, ε, ε, μιλώντας για την ασφάλεια καταθέσεων, την οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσει ε, το Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να ρωτήσω για την μεταρρύθμιση του ESM, διότι δεν έχει ακόμα επιληθεί το θέμα της δυνατότητας να υπάρχει κάποια ρευστότητα ή κάποια διευκόλυνση ρευστότητας ως τελευταία ή ε, στα τη λύση. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας για τις συζητήσεις όπως εξελίσσονται στο Συμβούλιο. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, δόθη εντολή στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ε, να εκπονήσει μια θέση ως προς το ενδεχόμενο να αφαιρείται από το κεφάλαιο ε, οι επενδύσεις σε software. Ε, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το software, ε, το λογισμικό των τραπεζικών ε, ε, ιδρυμάτων θα μπορεί να αποτελέσει κεφάλαιο σε περίπτωση εξυγίανσης ε, και αν μπορεί να θεωρείται λογιστικό αγαθό σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση ε, του νομισματικού συστήματος είναι κάτι που το παρακολουθούμε. Δεν συμμετέχουμε, δεν έχουμε λόγο. Έχουμε συμβάλει στο να είναι το ESM σαν πάροχος του δικτύου ασφαλείας. Διστάζουν τα κράτη-μέλη να κάνουν το ESM πάροχο ρευστότητας. Δεν συμμετέχουμε στο ESM. Αλλά εδώ εκφράζουμε άποψη και σταματάμε. Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε πλήρω. Η δεύτερη ερώτηση είναι λεπτομερέστατη. Μέχρι τώρα, για σχεδιασμό εξυγένση, πάντα βασιστήκαμε στην, στον ορισμό του κεφαλαίου το συνετό. Όταν χρειάζεται επανακεφαλοποίηση, θα πρέπει βάσει τη συνετή διαχείριση να κινηθεί κανεί. Κάποια στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται σαν στοιχείο ενεργητικού που θα μπορεί να υλοποιηθεί και να απολυθεί στα πλαίσια εξυγίανσης. Εδώ είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να γεφυρώσουμε τις στοιχές της ανάκαμψης που δεν είναι τόσο λογισμικό αλλά για θυγατρικές μπορεί να γίνει υλοποίηση των στοιχείων ενεργητικού στα πλαίσια εξυγίανσης αν δεν το χρησιμοποιήσει στην περίοδο ανάκτησης, μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην περίοδο εξυγίανσης. Ξεκινάμε από τον ορισμό της συνετής διαχείρισης και η όλη συζήτηση και οι λεπτομέρειες αφορούν τον εποπτικό φορέα. Ευχαριστώ. Ένα σημείο είναι σημαντικό. Αναφερθήκατε στο ESM και το backstop, το δίκτυο ασφαλείας. Το σχέδιο του, της συνθήκης απετέλεσε αντικείμενο συμφωνίας στο Eurogroup. Εξαρτάται το backstop με την μη τροποποίηση της μονιμότητας του νομικού πλαισίου για την εξυγένση των τραπεζών. Είναι σωστή η γενική αρχή, αλλά δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως νομικός περιορισμός όσον αφορά τα προνόμιο των συνομοθετών σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία εάν είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το πλαίσιο. Η δεμή θα υπήρχε περιορισμό ομοφωνία για μια συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία για το σχετικό μηχανισμό. Αυτό για να δείξουμε ότι πολιτικός πώς είναι σημαντικό. Χρειάζεται εξισορρόπηση επιμερισμού κινδύνου και μειώσεις του κινδύνου. Χρειάζονται εξέταση νομικές λεπτομέρειες να υπάρχει σωστή αντίληψη του θέματος και να εισακουστεί το Κοινοβούλιο στον αφορά τα προνόμια. Κύριος Κάριγκαμ, ευχαριστώ. Κυρία Κένιγκ, ερώτηση για τη ρευστότητα μετά την εξυγίανση. Είναι το πιο επικίνδυνο κενό που υφίσταται στο σύστημα σε περίπτωση ενδεχομένου πανικού. Ιούνιος 2017 η Banco Popular είπατε ότι ήταν επιτυχία. Η τράπεζα από μία ώρα ε, πριν ανοίξει τις πόρτες της βρέθηκε όταν λήφθη η απόφαση Αντάντερ να εξαγοράσει την τράπεζα για ένα ευρώ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να συμβεί αν η Σανταντέρ στο τέλος είπε δεν θέλουμε να την αγοράσουμε. Θα βλέπαν παιχνίδι τόλμης μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρών. Ποιο θα δηλιάσει πρώτο. Δεν ξέρω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ερώτηση. Αν πάμε δύο χρόνια μετά, Τετάρτη Ιουλίου, Ιουνίου, Ιουλίου, και είχαμε μεσαία, ή μεγάλο φορέα, μεσαίο μεγάλο φορέα, με 140 δις ή παρόμοιο μέγεθος τέλο πάντων. Έχουμε προχωρήσει για να αποφύγουμε ενδεχόμενο πανικό. Εάν όχι, Αναμένετε κάτι παρόμοιο. Εάν δεν βρεθεί λύση την τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει εργαλείο για παροχή ρευστότητα. Και αν αυτό ισχύει, τι προβλέπετε. Τι θα κάνατε. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να το αποφύγουμε αυτό. Υπάρχει ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή το οποίο ισχύει για όλη την Τραπεζική Ένωση και στην ουσία για όλη την Ευρώπη και είναι το λεγόμενο εργαλείο moratorium, το οποίο μας δίνει δύο ημέρες χρόνο. Τώρα αρκεί αυτός ο χρόνος, όχι. Βοηθά όμως, διότι για την περίπτωση της Banco Popular δεν υπήρχε moratorium των δύο ημερών, επομένως έπρεπε να βρεθεί μια λύση για να μπορέσει να ξανανοίξει η τράπεζα την Τετάρτη. Ε, ισχύει όμως τώρα πια, είναι ένα moratorium δύο ημερών, ε, είναι κάτι παραπάνω από το τίποτα που είχαμε πριν, επομένως είναι ένα πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι ότι έκτοτε ε, υπάρχει μια συζήτηση διότι όλοι μας νομίζω το FSP, η Ευρώπη ε, δρούν βάσει τη προπόθεση ότι κεφαλαιοποιεί την τράπεζα και θα υπάρξει ρευστότητα. Η ρευστότητα όμω δεν έρχεται μια ανοιχτή την επομένη. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το ξανακάνουμε τρίτη, αλλά λέμε συνεχώς ότι χρειάζεται μια λύση για τη ρευστότητα ε, στην εξυγίανση. Έχουμε προσφέρει μια λύση η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ε, μία εγγύηση για τις πρώτες απώλειες του ESRB και από εκεί και πέρα κάποια περαιτέρω βήματα. Αλλά εν τέλει για να έχουμε ρευστότητα το μεγαλύτερο ποσό ε, πολύ γρήγορα, ώστε να πείσει και αυτούς που έχουν προβλήματα, πρέπει να προέρχεται από τις κεντρικές τράπεζες και πρέπει να είμαστε ε, βέβαιοι ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν θα δώσουν ε, ρευστότητα χωρίς ε, εγγύηση. Επομένως, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι άνθρωπος αισιόδοξο, αλλιώ δεν θα είχα λάβει ποτέ αυτή τη θέση. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο όμως ε, προέρχεται με εγγύηση από το ε, Ταμείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα αντίστοιχο σύστημα το οποίο προέρχεται με εγγύηση από το Treasury των Ηνωμένων αλλά και εμεί χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο. Όπω λέω, αν χρειαστεί πάντα θα βρούμε μια λύση, αλλά δεν θέλω ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε το moratorium συνεχώ. Μα δίνει όμω τουλάχιστον αυτό το περιφέρειο δύο μερών για να λύσουμε το πρόβλημα. Νομίζω έχω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχουμε λίγο χρόνο, είναι το θέμα της συμμετρίας ε, στην εξυγίεση με τη ρευστοποίηση. Ε, το πρόβλημα με αυτό που συνέβη το 2017 και με τις Ιταλικές τράπεζες λίγο αργότερα ε, έθεσε θέμα ασφάλειας δικαίου. Τι θα γίνει αν εξετάσουμε την κάθε τράπεζα αναπερίπτωση, να θεωρήσουμε δηλαδή μια τράπεζα επαρκώς σημαντική για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει κάποιο κριτήριο, δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο κριτήριο. Πρόσφατα, ελπίζω τουλάχιστον, ε, αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας ή στις επόμενες ημέρες θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν είμαι βέβαιη γιατί το έχω υπογράψει αλλά δεν έλεγξα. Ε, ε, τι σημαίνει ενδιαφέρον δημοσίου συμφέροντος. Γνέφεται καταφωτικά, άρα υπάρχει στην ιστοσελίδα. Στην ουσία αυτό είναι μία απόπειρα να εξηγήσει λίγο κάπως αυτό το πλαίσιο αλλά το δεύτερο βήμα είναι αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Όταν αναφερόμαστε σε ρευστοποίηση, ε, εθνική διαδικασία φυραγγιότητας, ε, έχουμε 19 διαφορετικές διαδικασίες. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο βήμα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ελπίζουμε, για τη ρευστοποίηση των τραπεζών. Και ελπίζουμε και καλό πλαίσιο, λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίως. Ελπίζω να μην χρησιμοποιούμε το μανατόριο των δύο ημερών ε, αν υπάρχει κρίση για να βρούμε λύση για τη ρευστοποίηση. Καλύτερα αυτά να τα γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Σε περίπτωση ανάγκης ελπίζω να βρούμε μία λύση εκτάκτου ανάγκης. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε μια λύση ε, που θα κάνει καταμερισμό των κερδών. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια λύση. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ο Ερνές Ουρτασούν. Σβέν, ο κύριος Γκίγκολτ. Καταρχάς να σας καλωσορίσω από τους Πρασίνους ε, επί, ε, επίσης και θα ήθελα να κάνω μια πρώτη ερώτηση για να δώσω συνέχεια στην ερώτηση του Μάρκου Φέρμπερ όσον αφορά την κατάσταση των σχεδίων εξυγίανσης. Και πιο συγκεκριμένα υπήρξαν επικρίσεις ε, από, από το ελεγκτικό συνέδριο ε, λένε ότι δεν υπάρχουν και σαφείς δηλώσεις για το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα εξυγίασης ε, κάποιων τραπεζών. Μπορείτε να μας πείτε εσείς ε, για πόσες τράπεζες μπορείτε τώρα να πείτε στην τεκμηρίωσή σας ότι οι τράπεζες έχουν δυνατότητα εξυγίασης. Και δεύτερον, μπορείτε να δεσμευτείτε να μας στείλετε πιο αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση του σχεδιασμού εξυγίανσης και ε, που θα περιλαμβάνει και τα προσκόμματα τα οποία αντιμετωπίσατε λόγω του σχεδιασμού για την εξογήινση στη διαδικασία. Και δεύτερον, έχω και μία σύντομη ερώτηση σε συνέχεια της ετήσιας έκθεσής σας. Λέτε ότι όσον αφορά το Ταμείο, οι επιδόσεις και η επιτυχία στις επενδύσεις είναι λίγο αμφίβολη. Όσον αφορά τις εγγυήσεις, λοιπόν, έχετε μείον 0,16% κέρδος και όσον αφορά τις επενδύσεις σε ρευστό είμαστε στο μείον 0,4% που ποθανώς είναι λόγω του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είστε ε, ικανοποιημένοι με την επιτυχία των επενδύσεων. Θα ζητούσατε από κάποιον, για παράδειγμα, από εσά να επενδύσει με τέτοιε επιδόσεις και τι θα μπορούσατε να κάνετε για να ε, βελτιώσετε την επιτυχία των επιδόσεων. Βλέπω ότι δεν είστε και πολύ ικανοποιημένοι με αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι κανείς ε, προς το παρόν όταν πρέπει να επενδύσει χρήματα και τα επενδύει όπως εμείς με τρόπο που ε, θα μπορούν να τα ρευστοποιήσουν εύκολα ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να έχουμε ρευστότητα ε, δεν είναι δυνατόν να είναι επιτυχη... Ε, ικανοποιημένος. παρακολουθούμε την νομισματική πολιτική. Έχουμε το 0,4% σε λογαριασμούς ρευστού σε κεντρικές τράπεζες και συζητούμε και με το τμήμα προγραμματισμού που έχει ρόλο και στη στρατηγική επενδύσεων για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσουμε. Αν δείτε κάποια από τα στοιχεία ενεργητικού, το μείον 0,4 μια χαρά φαίνεται. Προσπαθούμε λοιπόν πολύ προσεκτικά να επενδύσουμε Έχουμε ένα πολύ περιορισμένο χαρτοφυλάκιο και παρεμπιπτόντω έχουμε κάνει εξωτερική ανάθεση. Προσπαθούμε να βρούμε τώρα και ένα δεύτερο εταίρο στον οποίο θα κάνουμε εξωτερική ανάθεση. Ε, τώρα, αν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τι επιδόσει, νομίζω ότι αυτό ε, είναι κάτι που ε, συμμεριζόμαστε με όλου εκείνου εδώ στην αίθουσα που προσπαθούν να επενδύσουν χρήματα και να συνεχίσουν να έχουν ρευστότητα. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη, αλλά νομίζω ότι η ομάδα μα έκανε καλή δουλειά. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη, την πρώτη σα ερώτηση, την κατάσταση κατάσταση των σχεδίων δεν έχουμε ολοκληρώσει κανένα πρόγραμμα εξυγίανσης με χαμόγελο λέγοντας ότι αυτή η τράπεζα μπορεί να διασωθεί. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα AMREL, ε, να υπάρχουν βασικοί ειδηπόροι και κάποια στοιχεία ενεργητικού. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν ε, υπάρχει ένα σχέδιο, πώς θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμόσει η Εθνική Αρχή την απόφαση. Υπάρχει λοιπόν ακόμα πολλή δουλειά. Ε, υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, επιχειρησιακή συνέχεια, ο ορισμός, ε, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται σταδιακά, σιγά σιγά, είναι δουλειά σε εξέλιξη. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει καλά σε κάποιους τομείς, κάπου αλλού πηγαίνουμε λίγο πιο αργά και... Ε, θέλουμε να δημοσιεύσουμε αυτές τις λεγόμενες προσδοκίες των τραπεζών, expectations to banks όπως τις αποκαλούμε, για να έχουμε ένα σαφές ετήσιο χρονοδιάγραμμα για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. Τώρα, αν είμαστε διατεθειμένοι να σας στείλουμε περισσότερα, εάν στείλετε ερώτηση, πολύ ευχαρίστω να αποπειραθούμε να απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με διάφορα χαρακτηριστικά ε, διάσωσης. Ευχαριστώ. Ο Γκούναρ Μπέκ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αρχές του έτους Μιλήσατε για φόβο επειδή το Brexit θα μπορούσε να αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τέλη Μαρτίου ξεκαθαρίσατε ότι βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιες ε, αλλαγές και κλειδονισμοί στις τιμές. Εξ όσων θυμάμαι είχατε ζητήσει μία παράταση από το Συμβουλίο του άρθρου 50 Λοιπόν, πριν την παρέτηση της κυρίας Μέη, έχω να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η αρχική σας τοποθέτηση ότι το Brexit δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι αντίθεση με... είναι αντίθετη, με συγχωρείτε, με τις δηλώσεις του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν του κυρίου Ντομπρόφσκης ε, στις Απριλίου και του κυρίου Ντράκη της 10 Απριλίου και οι δύο μίλησαν για πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις μιας κρίσης ρευστότητας σε συνδυασμό με τον Brexit. κάτι το οποίο θα καθιστούσε αναγκαία μια επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης τη Τράπεζα, Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πώς αξιολογείτε αυτές τις διαφορές εκτός αν οι κύριοι Ντομπρόφσκης και Ντράγκη απλά αναζητούν προσχήματα για περισσότερη ποσοτική χαλάρωση. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Η εκτίμησή σας για τους κινδύνους του Brexit για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα υπό, πως έχει αλλάξει υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων. Αναφέρομαι στην καθυστέρηση του Brexit Μιλάμε για 31 Οκτωβρίου ή και παραπέρα για την παρέτηση της κυρίας Μέη και την πιθανή διαδοχή της από τον Μπόρις Τζόνσον στην Πρωθυπουργία. Να προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας σύντομα. Το σχόλιο μου αφορούσε τη δουλειά που κάναμε εμείς έτσι ώστε οι τράπεζες να είναι σε θέση να εξηγιανθούν και το τι θα σήμαινε το Brexit για τις τράπεζες. Οπότε στα τέλη του προηγούμενου έτους, τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο, ήμασταν έτοιμοι να πούμε ότι θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τις ε, τράπεζες, να έχουν εκδώσει ομόλογα ε, υπό αγγλικό δικαίωμα που έχουν κάνει πολλές και ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Brexit ε, ίσως αυτά να μην ε, θεωρούνται πλέον μέσω MRL. Δεύτερον, συνεργαστήκαμε στενά με τις υποπτικές αρχές ε, για να πούμε ότι όταν οι τράπεζες θα πρέπει να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τι αναμένουμε εμείς από τη σκοπιά της δυνατότητας εξυγίανσης, οπότε να μην είναι δηλαδή γραμματοκιβώτιο κτλ να μεταφερθούν κανονικά. Αυτά τα βάλαμε στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, αν με ρωτάτε αν είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι, όπως με είχαν ρωτήσει, είχα πει ότι είμαστε όσο προετοιμασμένοι γίνεται. Δεν είναι μυστικό ότι σαφώς με την αναβολή του Brexit κάποιες από τις δραστηριότητες που είχαν προγραμματίσει οι τράπεζες επιβραδύνθηκαν κάπως, οπότε το μήνυμά μου σήμερα στις τράπεζες είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να το αναβάλουν, πρέπει να είναι έτοιμες, να οργανωθούν και το συμπέρασμα στο οποίο επιμένω είναι ότι δεν βλέπω κάποιον άμεσο κίνδυνο. Εξακολουθεί να ισχύει, αλλά πάντα αυτό το έλεγα μαζί με κάτι άλλο, ότι κάποια δευτερογενή αποτελέσματα από την οικονομική επιβράδυνση που θα προκαλέσει το Brexit είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε. Αλλά οι χρηματαγορές ίσως να μην είναι η αφορμή, ίσως αυτό να, να είναι κάποιες δευτερογενείς επιπτώσεις. Και αυτό δεν είναι αντιφατικό με τα όσα είπαν οι κύριοι Ντομπρόφσκη και Ντράγκη. Σας ευχαριστώ. Ντέρκ Γιάν Έπινγκ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς την κυρία Κένιχ και αφορά την Deutsche Bank, η οποία σήμερα κάνει μια τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια για να βγει από την κρίση ε, ε, με το σχέδιο αυτό το φιλόδοξο που λέγεται Καΐρο, δεν ξέρω γιατί το λένε έτσι. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξής. Όταν μπαίνετε σε τέτοια προβλήματα, μιλάμε για κάποια κρίση, για χρεοκοπία. Και δεύτερον, όταν μια τράπεζα τέτοιου μεγέθους ε, περνάει σε μια τέτοια διαδικασία, τι ε, μπορείτε να κάνετε, γιατί τα κονδύλια σας είναι μόνο 33 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση. Κοιτάξτε, ε, είναι κανόνας ότι δεν σχολιάζω συγκεκριμένα ε, πιστοτικά ιδρύματα, αλλά μια που η Deutsche Bank είναι μια παγκόσμια συστημική τράπεζα, κάνουμε σχέδια εξυγίανσης και θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Μάρκους Φέρμπερ, ελπίζω να μην χρειαστεί να εξυγιάνουμε πολλές τράπεζες ελπίζω να υπάρχουν σχέδια ώστε να λύσουν τα προβλήματά τους μόνες τους. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο εξυγένσης βεβαίως για την Deutsche Bank. Υπάρχουν οι απαιτήσει MRL και τα σχετικά και θα μείνω σε αυτά. Εάν μια τράπεζα αρμοδιότητός μας ε, χρεοκοπείται, έχουμε μια ε, σειρά εργαλείων. Έχουμε παραδείγματος χάρη την πώληση δραστηριοτήτων, όπως στην περίπτωση της Banco Popular, όπου ήμασταν τυχεροί, υπήρχε αγοραστής ενδιαφερόμενος για να αγοράσει τις δραστηριότητες. Το εναλλακτικό σενάριο είναι ότι στην περίπτωση αυτή θα ξεκαθαρίσουμε τις ζημιές και θα ανακεφαλαιοποιήσουμε κάνοντας το MREL κεφάλαιο. Αυτό το οποίο λέμε δηλαδή ε, ένα ανοιχτό bail-in ε, τραπεζών. Αυτές είναι βασικά οι επιλογές. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλά αυτό αποδεικνύει ότι το Emerald είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σου δίνει επιλογές στο τι μπορείς να κάνεις. Σας ευχαριστώ. Να έχετε και χρόνο για άλλη ερώτηση αν θέλετε. Ωραία, ευχαριστώ. Μάρτιν Σίρντεβαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Κένιχ. Εδώ είμαι. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ και μας ενημερώνετε για τις εργασίες του ΣΕΡΜΠΕΚ και για την ετήσια έκθεση. Αναφέρατε και αναφέρθηκαν και κάποιες ερωτήσεις στο ότι η εφαρμογή των μέσων εξυγίανσης ειδικά σε κάποιες μεγάλες τράπεζες καθυστερεί. Θα ήθελα να γνωρίζω ε, πώς εκτιμά την κατάσταση, γιατί συμβαίνει αυτό και εάν αυτό πιθανώς θα έχει κάποιες συνέπειες για την σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Δέκα χρόνια μετά την τραπεζική κρίση μας λέτε πως ε, θα πρέπει να αποφευχθεί ένα ακόμα bailout. Και δεν ξέρω αν είμαστε σε τέτοια θέση. Και άλλη μια ερώτηση σε σχέση με την ετήσια έκθεσή σας. Λέτε ότι θα πρέπει οι τράπεζες να είναι σε θέση να εξηγιανθούν όμως η περιπλοκότητα κάποιων τραπεζικών ομίλων δυσκολεύει ακριβώς ε, αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε το ESRB να παίξει έναν σημαντικότερο ρόλο για να μειώσει την περιπλοκότητα αυτή και να υπάρχει δυνατότητα εξυγένσης και μια τρίτη σύντομη ερώτηση και αυτό αναφέρθηκε δεν έχετε ακόμα στελεχωθεί πλήρως γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Ε, λογικό θα ήταν να ε, έχετε πλήρη στελέχωση για να μπορέσετε να σταθεροποιήσετε τον τραπεζικό τομέα. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας. Να ξεκινήσω με την τελευταία σας ερώτηση για τη στελέχωση. Ε, βρισκόμαστε σε μια ανταγωνιστική αγορά, τα έχω πει και την προηγούμενη φορά, ήμασταν τυχεροί που Είχαμε ανθρώπους από τις τράπεζες, από τις εποπτικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά χρειάζεται χρόνος, είναι μια διαδικασία μακροσκελής και δυστυχώς φέτος ε, χάσαμε σε διαγωνισμό, στον ανταγωνισμό αν θέλετε ε, προσωπικό από την Κομισιόν που αναζητούσε προσωπικό και ε, δυστυχώς το προσωπικό μου ήταν τόσο καλό ώστε τους έγιναν προσφορές και επέλεξαν να πάνε στην Κομισιόν. Οπότε... Εντάξει, θα ήμουν και δυστυχής εάν δεν έπαιρναν το δικό μας προσωπικό, γιατί είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Αλλά είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δεύτερον, για τον δικό μας ε, τον ρόλο. Νομίζω ότι έχω παρεξηγηθεί κάπως όταν λέω ότι οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγενθούν. Ε, δεν είναι ότι δεν έχουμε φιλοδοξία, αλλά θεωρώ ότι ε, το να δείχνουμε κάτι και να λέμε η δομή αυτή είναι πολύ πολύ πλοκή και δεν θα λειτουργήσει, η απάντηση πρέπει να έρθει πρώτα από την τράπεζα και μετά θα αξιολογήσουμε αν είναι μια απάντηση ικανοποιητική ή όχι. Εμείς δεν είμαστε ο σύμβουλός τους, ε, για την δομή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις, αλλά η εφαρμογή. Τώρα όταν μιλάμε για δεδομένα είναι εύκολο να πούμε ότι πρέπει να γίνουν γρηγορότερα τα συστήματα πληροφορικής σας. Πρέπει να υπάρχουν δεδομένα με το πάτημα ένα σκουπιού. Εμείς το λέμε, αλλά πρέπει η τράπεζα να το κάνει. Εμείς λέμε γιατί δεν το κάνετε και αναλαμβάνουμε δράση. Τέλος, η εφαρμογή των μέτρων μας Μιλήσατε για καθυστέρηση και δισταγμούς. Δεν νομίζω. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί. Ε, δεν θέλουμε να προκαλέσουμε την κρίση την οποία θέλουμε να αποτρέψουμε. Μπορούμε να μιλάμε και να λέμε γρήγορα αυτό πρέπει να γίνει σε 6 μήνες, σε 9 μήνες, αλλά ρεαλιστικά οι τράπεζε χρειάζονται χρόνο να το εφαρμόσουν. Το ίδιο ισχύει και για τους στόχου MREL επίση. Πράγματι. Σας ευχαριστώ. Λίδια Περέιρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ κυρία Κένινγκ για την παρουσία σας εδώ. Κάποιες ερωτήσεις έχω σχετικά με αυτά που είπατε. Στόχο, στόχος μας η ολοκλήρωση της ε, Ένωσης των Κεφαλαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης. Βλέπουμε τώρα μια επιβράδυνση της οικονομίας. Αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα ακόμα όσον αφορά το κρατικό χρέος, κυρίως σε χώρες όπως η Ιταλία ή η Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά την έκθεση των χωρών αυτών και των τραπεζών αυτών στο κρατικό χρέος. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Σχετίζεται και με τη δυνατότητα εξήγησης των τραπεζών εν γέννη. Απάντηση. Προσπαθώ να μείνω στην περιοχή μου, στην αρμοδιότητά μου και το δημόσιο, το κρατικό χρέος δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Να πω κάτι ξεκάθαρο. Είδαμε δύο αρκετά καλά χρόνια και ακόμα καλή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει και τις τράπεζες. Μπορούν να θέσουν τα του οίκου τους εντάξει και να ετοιμαστούν για χαλεπούς καιρούς. Και εγκρίνουμε πλήρως τις δραστηριότητες που καταβάλλονται για να γίνουν οι σωστές κινήσεις. Και έτσι, αν γίνουν πιο δύσκολες οι καταστάσεις, να μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη αφετηρία. Ευχαριστώ. Θέλετε να υποβάλλετε και άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Μπίλι Γκάλαχερ. Ευχαριστώ, κυρία Κένιγκ. Δύο σημεία να θέσω. Έχω υπηρετήσει σε κυβέρνηση της Ιρλανδίας την οικονομική κρίση και όταν μιλάτε για κεφαλαγορές, bail-out και ρευστότητα, ανατριχιάζω. Δύο ερωτήσεις έχω. Τι σύστημα εγκαίρου προειδοποίησης υπάρχει όταν η τράμες, τράπεζα αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Διότι πολύ γρήγορα το πρόβλημα ρευστότητας γίνεται πρόβλημα κεφαλουχικό, αν δεν λυθεί γρήγορα αν είναι συστημικά σημαντική μια τράπεζα. Τι μηχανισμοί υπάρχουν για να εντοπιστεί το πρόβλημα πριν έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα αργά το βράδυ ή στην πόρτα της εθνικής κυβερνήσεως αργά το βράδυ ε, ζητώντας βοήθεια όπως έγινε στην Ιρλανδία αλλά και αλλού στην Ευρωζώνη το 2010. Άλλο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τη συνετή διαχείριση του νομίσματος ε, της Ευρωζώνης, αλλά εντός αυτού του πλαισίου μου δημιουργείται μια ανησυχία. Υπάρχουν υποχρεώσεις συνετής διαχείρισης που δύσκολα αντιμετωπίζουν προβλήματα εντός τραπεζών. Κυρίως ε, η αφαίρεση κέρδους ε, από τους πελάτες. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην Ευρωζώνη με τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόσβαση στην δανειοδότηση είναι διαφοροποιημένη με άλλα λόγια. Έχετε άποψη πάνω σε αυτό. Ε, πάντα εγώ έχω κάποιες υπόνοιες ότι όταν έχουν προβλήματα οι τράπεζες αφαιρούν τα κέρδη από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους κατόχους ε, στεγαστικών δανείων. Απάντηση. Είναι ένα θέμα για το SSM και όχι για μας. Δεν θέλω να σχολιάσω. Σύστημα εγκαίρου προειδοποίησης υπάρχει. Ομολογώ ότι πράγματι οι κρίσεις ρευστότητας μπορεί να εξελιχθούν τάχιστα σε κάποιες περιπτώσεις. Μία κρίση ρευστότητας είναι γενεσιουργός μάλλον προκαλείται από πρόβλημα αφαιρεγκαιότητας και από άλλους λόγους. Το σύστημα εγκαίρου προειδοποίησεως που υπάρχει είναι συνδυασμός συστήματος εγκαίρου προειδοποίησεως που χρησιμοποιεί το SSM. Έχουμε πλήρη ευθεγράμμιση με το SSM για οιασδήποτε τράπεζε που έχουν πρόβλημα και συνεργαζόμαστε. Παρακολουθούν οι ομάδε μα τι τράπεζες. Δεν θα είναι ρεαλιστικό να πω ότι ποτέ δεν θα εκπλαγούμε Χρειάζεται πρόληψη, πρόνοια, να παρακολουθούμε το σύστημα, να το ελέγχουμε αρκετά, ούτως ώστε πάντα να υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση ε, σε αρκετό χρονικό διάστημα πριν ξεσπάσει η κρίση. Στα πλαίσια των τραπεζών που δεν έχουν ισοζύγιο στον προπολογισμό τους. Αν μιλάμε για την Τραπεζική Ένωση την Ενία αγορά, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εργάζονται σωστά οι πολίτε. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό εκεί που δεν υπάρχει. Το είπε και ο Μάριο Ντράγκη. Σχεδόν μονοπόλιο επικρατεί στην Ιρλανδία από πλευρά τραπεζική. Όταν μιλάμε για τραπεζική ένωση, δεν θα πρέπει να πλήττονται οι ε, πολίτες μιας χώρας αν δεν έχουν τα επιτόκια μπορούν να έχουν στη Γαλλία, στην Γερμανία ή στην Πορτογαλία οι Ιρλανδοί. Μπορούν να υπάρξουν μέτρα που θα επιβληθούν σε τράπεζες οι οποίες δεν ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες της ανοιχτής αγοράς και τελικά δεν υλοποιείται η πραγματική ενιαία αγορά που αφορά τους πολίτες. Ευρύτατο το ερώτημα, είναι η απάντηση. Τίθεται και το θέμα αν ε, βλέπουμε δεσυνορικές δραστηριότητε ή κινούνται σε πολύ τοπικό επίπεδο οι τράπεζες. Νομίζω κινούνται σε τοπικό επίπεδο πολύ οι ε, τράπεζες. Αυτό δεν αφορά την αρχή για την διάσωση. Εμείς σαν θεματοφύλακα θέλουμε να φροντίσουμε να βρούμε απάντηση αν κάποια τράπεζα έχει προβλήματα οικονομικά. Πώς προστατεύουμε τους κατόχους ομολόγων, τους φορολογούμενους, όχι τους μετόχους, τους καταθέτες από τον αντίκτυπο αυτού. Αλλά συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα, αλλά είναι περισσότερο συνδυασμός ενό συσκεφαλογορών θέμα εποπτείας και ίσως συμπεριφοράς και συνηθιών. Ευχαριστώ. Η Ορόλα Λουκ, συγγνώμη που άλλαξα τη σειρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρία μου. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Μιλήσαμε για την οικονομική επικαιρότητα που ε, έχει στο προσκήνιο την Deutsche Bank και η Deutsche Bank διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και το παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι η μόνη, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ε, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 τις συνέπειες ε, του σκιώδους τραπεζικού τραπεζικού συστήματος για την ποιότητα. Ξέρουμε ότι ήταν περίπλοκο και για τους ρυθμιστές για να δουν επακριβώς τι συμβαίνει σε αυτό το παράλληλο τραπεζικό σύστημα και το 2007 εκτιμόταν ότι ήταν 52 δις οι δραστηριότητες, 52 δις δολάρια, ε, ένα ποσό το οποίο αυξανόταν συνεχώς κυρίως στην Ευρώπη. Πλέον έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο κάνει νομισματική δημιουργία χωρίς να πρέπει ε, να ε, εξαρτάται από τις τράπεζες που κάνουν τη νομισματική δημιουργία. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος ρευστότητας και τελικά και ένα συστημικός κίνδυνος ο οποίος ε, τίθεται ακριβώς από αυτό το σκιώδε τραπεζικό σύστημα. Η ερώτηση μου είναι αν μπορείτε να κάνετε σωστά την αποστολή σας χωρίς να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία του ε, παράλληλου τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει μία δέσμη μέτρων για τις τράπεζε, μήπω θα έπρεπε να έχουμε και μία δέσμη μέτρων ε, για αυτές τις μορφές ε, ε, συναλλαγών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σύστημα. Τι κάνετε εσείς για να αντιμετωπίσετε όλη αυτή τη σκιώδη κατάσταση και ε, μήπως για να μπορέσετε να εκτελέσετε σωστά την αποστολή σας ε, θα έπρεπε να υπάρχει και μια νομοθετική πρόταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση του παράλληλου τραπεζικού συστήματος. το σκιώδες ε, τραπεζικό σύστημα είναι κάτι το οποίο γνώριζα στην προηγούμενη ε, επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αν είναι ο κίνδυνο ο ίδιο, θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνε. Επομένω, πρόκειται για σαφέ ζήτημα. Αλλά σίγουρα ε, δεν είναι θέμα το οποίο απασχολεί το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανση. Εμεί εξετάζουμε την ε, σύνδεση των αγορών και θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε τον κάθε κίνδυνο και από αυτή την οπτική σκοπιά, αν υπάρχουν δυνατότητες για ρευστότητα και ούτω καθεξής. Αλλά ο βασικός ε, στόχος της διασύνδεσης δεν είναι προς το παρόν ο κίνδυνος από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, είναι κάτι το οποίο ανέφερα πολύ σύντομα, η κεντρική αντισυμβαλόμενη, όπου η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρωζώνης ή μάλλον και η μεγαλύτερη τράπεζα παγκοσμίω, είναι και ε, το βασικό, ο βασικός ε, ε, υπεύθυνο εκαθάριση. Εάν αποτύχει λοιπόν ε, ένα εξ αυτών, θα έχουμε και ένα φαινόμενο ντόμινο στο σύστημα. Το Κοινοβούλιο ξεκίνησε ε, τις συζητήσεις για το EFSP2 και ε, τις αποφάσεις, τα rulings και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε. Έχετε δίκιο ο Μάρκος Φέρμπερ. Ähm, Ευχαριστώ. Με το τραπεζικό πακέτο έγινε μια εισαγωγή στις ε, υποχρεώσεις δημοσιότητας για τα έμπρελ και τα σχετικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσαν ε, ασθενέστερα πιστοτικά ιδρύματα να βρεθούν σε δυσκολότερη θέση. Στη ΣΥΠΑ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κατόφλια όσον αφορά τις υποχρεώσεις ε, δημοσιότητας για τις δυνατότητες εξυγένσης και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής ε, Σταθερότητας έκανε προσφάτως μια σχετική διαβούλευση. Θα ήθελα να μας κάνετε μια εκτίμηση της κατάστασης αυτής εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι υπάρχουν μειονεκτήματα όσον αφορά την δημοσιότητα σχεδίων εξυγίανση ε, και ποια κομμάτια θεωρείτε ότι θα έπρεπε να δημοσιεύονται και ποια όχι. Α, δύσκολη ερώτηση. Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Όπο, ναι. Έμπλεξα και τις γλώσσες. Συνήθως προσπαθώ να μιλώ αγγλικά. Ε. I fully agree that we should... Συμφωνώ ότι σταδιακά θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για το κατά πόσον μπορεί να εξηγενθεί μια τράπεζα. Αλλά αυτή είναι άσκηση ισορροπίας. Ε, εάν δημοσιεύσει το σχέδιο εξυγιανθεί, ελοχεύει και ο κίνδυνος οι αγορές να ε, πιστέψουν ότι αυτό θα συμβεί και ξέρουμε ότι γίνεται ένα πρώτο σχέδιο, ένα δεύτερο σχέδιο και μετά μπορεί η πραγματικότητα να ε, έρθει να χτυπήσει στο πιο αδύναμο σημείο της ε, δυνατότητας εξοικίασης. Νομίζω η Τράπεζα της Αγγλίας είπε πρόσφατα ότι εξετάζουν ε, να κάνουν αξιολόγηση κατά πόσον μπορούν να διασωθούν οι τράπεζες ή όχι και να τα δημοσιεύσουν ε, σταδιακά. Εγώ είμαι λίγο ουδέτερη. Είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και πώς θα πάει, διότι πριν από ένα χρόνο περίπου, ίσως και λίγο περισσότερο, ο Ελβετός ρυθμιστής δημοσίευσε στοιχεία και λέει ότι από τις χαμηλότερες, τις υψηλότερες απαιτήσει αφαίρεσαν ένα ε, ποσοστό ε, διότι οι τράπεζες θεωρήθηκε ότι έχουν αρκετή δυνατότητα εξυγίασης για να μπορέσουν να λάβουν κάτι περισσότερο. Και εγώ Περίμενα με ενδιαφέρον τι αντιδράσει. δεν είδα κάποια αντίδραση. Τους ε, κάλεσα και μου είπαν ότι ήταν μηδενική αντίδραση, δεν αντέδρασε κανεί. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά τα MRL, πάντα λέω ότι οι τράπεζε θα πρέπει να τα δημοσιεύουν, γιατί οι επενδυτές πρέπει να ξέρουν και πού επενδύουν. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε. Προς το παρόν διατηρώ ουδέτερη στάση. Ευχαριστώ. Έρωχε ένα ελώμα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Κιόνιν για αυτή την ε, πληρέστατη παρουσίαση. Έχουμε πλέον ε, τέσσερα χρόνια εμπειρίας και γι' αυτό ακριβώς ε, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις ώστε να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Πρώτον, συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων και του Συμβουλίου και με άλλα διεθνή ιδρύματα. Γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο κάνετε απαιτεί ε, πολύ ε, διεξοδική συνεργασία ώστε να μπορέσουν ε, να πάνε τα πάντα σωστά. Και εδώ έρχομαι και στην ερώτησή μου. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων και διεθνών ιδρυμάτων είναι η βέλτιστη δυνατή. Είστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ε, ιδρυμάτων. Δεύτερη ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση για τη ρευστότητα. Πρόκειται για ουσιαστικό θέμα, το γνωρίζουμε όλοι. Και αναφέρατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσω θα μπορούσε εδώ να διαδραματίσει κάποιο ρόλο προκειμένου να μπορεί να εγγυηθεί ρευστότητα. Να είναι ο εγγυητή αυτή της ρευστότητα. Πώ βλέπετε λοιπόν εσεί αυτό το ρόλο για την ΕΚΤ πιο συγκεκριμένα. Θέλετε πραγματικά ή μάλλον πιστεύετε πραγματικά ότι θα μπορούσε να παρέμβει η ΕΚΤ για να εγγυηθεί τη ρευστότητα περισσότερο από όσο κάνει τώρα, για παράδειγμα στην περίπτωση των ε, securities. προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση. Η συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ, ε, του SSM, της ε, Κομισιόν, των Εθνικών Αρχών και των ε, Εθνικών Αρχών Εξυγίανσης, που είναι μέλος του Κεντρικού Μηχανισμού Εξυγίανσης, είναι κάτι το θετικό. Όταν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία είναι ένα πρόβλημα ίσως προσωπικό που πρέπει να επιληθεί αλλά το βασικό πλαίσιο λειτουργεί ικανοποιητικά και αν υπάρχει κάποια εξαίρεση αποδεικνύει τον κανόνα ε, η ρευστότητα και είμαι ικανοποιημένη για αυτήν γιατί νομίζω ότι είμαστε πλέον σε καλή τροχιά η ρευστότητα στην εξυγένση σωστά επισημάνατε ότι παίρνουν να παίξουν το ρόλο οι κεντρικές τράπεζες, αλλά βεβαίως και το Συμβούλιο Συστημικής ε, Σταθερότητας, αλλά περιορισμένο. Όταν μιλάμε για την ρευστότητα και τις ανάγκες ρευστότητας μιας παγκοσμίω ε, συστημικής τράπεζας, μιλάμε για πολύ ικανό ποσό. Ε, το οποίο το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης πιθανότατα δεν θα επαρκεί αλλά το ενίο ταμείο εξυγένσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει εγγύηση στην κεντρική τράπεζα παραδείγματο χάρη. Και μετά το ερώτημα είναι πόσες εγγυήσει χρειάζονται, εάν είναι η πρώτη δόση κτλ. Η συζήτηση αυτή ε, είναι ένα εξελίξη αυτή τη στιγμή και όπως σας είπα είμαι αισιόδοξη Πάντα θεωρώ ότι θα βρεθεί μια λογική λύση, αλλά ένα είναι σίγουρο, το ταμείο αυτό ή το ταμείο συν το backstop δεν θα είναι η μόνη λύση. Δεν είναι ε, λεφτά χωρίς τέλος ε, και μιλάμε και για αριστότα η οποία θα πρέπει να είναι χαμηλού κινδύνου γιατί ε, θα πρέπει να έχουμε τελικά μια τράψα η οποία θα, είναι, ε, θα έχει εξηγιανθεί και θα είναι ανακεφαλαιοποιημένη. Οπότε η έκθεση θα πρέπει να είναι περιορισμένη. Σας ευχαριστώ, Ερνέστ Ουρτασούν. Ευχαριστώ, κυρία Κένικ, για να επανέλθω στα σχέδια εξυγίανσης. Ε, έχω αντιληφθεί ότι για να ολοκληρωθούν τα σχέδια αυτά είναι νομική απέτηση να γίνεται μια αξιολόγηση των ηχών εμποδίων της ε, δυνατότητας εξυγένσης. Θα ήθελα κάποιες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις από εσάς. Αυτές οι αξιολογήσεις έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, γίνονται ή όχι, ε, είναι ολοκληρωμένες και έχουμε ήδη αναπτύξει ή αφαιρέσει εμπόδια στην ικανότητα εξυγένσης από τα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκείνα στα οποία έχει γίνει η εξήγηση. Αλλιώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, ε, επίση από την ετήσια έκθεσή σα, λέτε ότι η μεθοδολογία για τράπεζες ε, οι οποίες ε, είναι στα όρια της χρεοκοπίας ε, ολοκληρώνεται. Αυτό είναι θετικό γιατί η μεθοδολογία αυτή ήταν κάτι το επίμαχο στο παρελθόν και θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ αυτής τη μεθοδολογία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με το δεύτερο ερώτημα. Έχουμε αναπτύξει την δική μα μεθοδολογία όπως ξέρετε έχουμε το ίδιο κατόφλι που έχει η ΕΚΤ για να καθορίσουμε πως μια τράπεζα κινδυνεύει αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η ΕΚΤ ως εποπτική αρχή ε, κατά μέσο όρο είναι πολύ πιο κοντά στην τράπεζα, έχει περισσότερες πληροφορίες, οπότε η δική μου η ανησυχία για την ώρα είναι να διασφαλίσουμε πως μία τράπεζα η οποία ε, βρίσκεται σε δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες για να λάβουμε μια απόφαση μόνοι μας. Ε, αυτά. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά στην δική μας μεθοδολογία και τη μεθοδολογία της ΕΚΤ. Πάντα είναι θέμα του να βρεθεί η ισορροπία για να μην δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα και βρεθούμε σε κάποιο κενό ή πολύ αργά. Εν ολίγης όμως η μεθοδολογία μας και η μεθοδολογία της ΕΚΤ είναι θα έλεγα συγκρίσιμες ε, και ισοδύναμες. Δεύτερη ερώτηση για τη δυνατότητα εξυγένσης. Έχω πει ότι... Να το επαναλάβω το κοιτάμε, έχουμε ε, κοιτάξει κάποια από αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν θα πω ότι ε, κάποια, οποιαδήποτε τράπεζα είναι εντάξει και μπορούμε να την ξεχάσουμε. Έχει δουλειά να γίνει σε όλες και όπως υποσχέθηκα και στον Σβεν Γκίγκολτ όταν στείλει ερωτήσεις θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε συγκεκριμένα στα διάφορα θέματα. Σας ευχαριστώ. Γκούναρ Μπέκ. Κύριε Πρόεδρε. Δείχνεται μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ότι μέσω του ταμείου σας θα μπορέσουν να εξηγιανθούν οι τράπεζες στο μέλλον χωρίς να προσφύγουν στο φορολογούμενο. Δεν είναι παραπλανητικό αυτό. Το SF χρηματοδοτείται από υποχρεωτικές εισφορές των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 3.100 τόσα το 2018. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εισφορών ε, κατ' ουσίαν, εφόσον το πληρώνουν οι τράπεζες, το πληρώνουν οι καταθέτες και οι επενδυτές ε, μέσω των ε, καταθεσιών τους. Άρα στην ανάγκη θα διασώσουν τράπεζες σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο δηλαδή το διαχωρίζει από ένα συνηθισμένο bailout είναι ότι τα λεφτά των φορολογουμένων περνάνε μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων των τραπεζών και αφαιρούνται εκ των προτέρων τράπεζες στην Βουλγαρία και στην Κροατία θα ενταχθούν στο Ταμείο τα επόμενα χρόνια. Και οι δύο αυτές χώρες έχουν πολύ ευπαθή τραπεζικό τομέα και τώρα θα έχουν δικαίωμα στήριξης. Η Βουλγαρία και η Κροατία έχουν και πολύ χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών που είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Οπότε ήδη εδώ πέρα δοκιμάζεται πολύ η λογική γιατί υπάρχει μια σχέση μεταξύ του χαμηλού ποσοστού αποταμίευσης και της πιθανότητας να χρειαστεί διάσωση μια τράπεζα, κάτι το οποίο εσείς διαψεύδετε. Παρόλα αυτά λοιπόν, και δεδομένων όλων αυτών μπορείτε εσείς ε, να πείσετε τους Γερμανούς αποταμιευτές και τους άλλους ότι ε, η φόβη μας είναι αδικαιολόγητη. Να προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας. Το ταμείο αυτό συστημικής σταθερότητα. Ε, χρηματοδοτείται από τον κλάδο. Βεβαίως ο κλάδος το χρηματοδοτεί από τα έσοδά του. Που σημαίνει ότι τα λεφτά είτε δεν πάνε στα κέρδη είτε ε, βγαίνουν από τις καθημερινές εργασίες τους. Αλλά το να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι από τα μιευτές ε, διασώζουν τις τράπεζες ε, απανταχού είναι κάπως τραβηγμένο. Και να λέμε μετά οι αποταμιευτές είναι φορολογούμενοι και αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Αναφέρεται τώρα και αυτό δεν το ανέφερα στην εισαγωγή μου, ότι πιθανώς ε, θα έχουμε δύο νέα μέλη της Τραπεζικής Ένωσης, την Βουλγαρία και την Κροατία. Θα πρέπει να δώσουν τα κονδύλια αυτά στο ενιαίο Ταμείο Εξυγένση όταν γίνουν μέλη και μην ξεχνάτε ότι μετά θα γίνει και ένα έλεγχο τη ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού τους και θα ε, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσει όπως κάθε μέλος. Αλλά το ενιαίο Ταμείο Εξυγένσης για εμάς είναι πάντα η τελευταία λύση. Οι τράπεζε πρέπει πρώτα να χρηματοδοτήσουν τις ζημίες από τους ε, μετόχους, ε, τους ομολογιούχους τους ε, και μετά ακολουθεί το ταμείο. Δι' δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι θα έχει υπάρξει ένα bail-in 8% των συνολικών ανοιγμάτων της τράπεζας που είναι αρκετά μεγάλο περιθώριο πριν υπάρχει πρόσβαση στο ταμείο. Σας ευχαριστώ. Φάμπιο Μάσιμο Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς κυρία Κένιγκ. Στην προηγούμενη θητεία, όπως υπενθυμίσατε και πριν, είχαμε πριν ψηφίσει το πακέτο τραπεζικό μαζί το Συμβούλιο και την αναθεώρηση που ε, καθόριζε τα θέματα αυτά, το Μπέιλιν και το Αμερέλ. Έχω κάποιες ερωτήσεις επ' αυτό. Η πρώτη ερώτηση. Έχετε πρόθεση να κάνετε μελέτες ποσοτικές, να δείτε τι αντίκτυπο έχουν οι απαιτήσει MRL στι διάφορες χώρες και στα διάφορα μοντέλα τραπεζών βάσει ε, των, των κειμένων της οδηγίας. Μετά που συνδέεται με κάποιες ε, μελέτες που έγιναν, κυρίως στη Bank Italia, ε, οι νέε απαιτήσει έχουν αντίκτυπο ασύμετρο στα διάφορα τραπεζικά συστήματα και στα διάφορα μοντέλα τα επιχειρηματικά με ενδεχόμενο αντίκτυπο αρνητικό όσον αφορά τη διαθεσιμότητα τη πίστοση. Πώ θα λάβετε υπόψη τέτοιε ενδεχόμενε αρνητικέ συνέπειε τη απαιτήσεω να γίνεται σεβαστή μια αρχή τη αναλογικότητα στον καθορισμό των MRL. Και θα ήθελα να ξέρω τι κάνετε με τον ρυσμό των στόχων MRL για τις τράπεζες σημαντικές, κυρίως πώς λαμβάνετε υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με την έκθεση σε ρευστοποιημένους και περίπλοκους τίτλους και την έκθεση εκτός του προπολογισμού των τραπεζών. Όπω σημειώνεται σε κάποιε τράπεζε, ε, κάποιε τράπεζε είναι εκτεθειμένε στα μέσα του επίπεδου 2 και 3, που είναι δύσκολο να αξιολογηθούν, άρα οι κίνδυνοι βαραίνουν, μάλλον ε, τελικά υποτιμούνται και κατά πολύ. Ευχαριστώ. Ο αντίκτυπος των αλλαγών του κανονισμού για τα διάφορα πεζικά μοντέλα για τις διάφορες χώρες είναι κάτι που θα αξιολογηθεί για την ώρα προσπαθούμε στην πολιτική μας να εφαρμόσουμε το νέο πακέτο. Συλλέγουμε για την ώρα στοιχεία για υπολογισμό MRL ετησίως. Και όπως κάναμε και το 2018 όταν δημοσιεύσαμε και την πολιτική μας, κάνουμε και αξιολόγηση αντικτύπου για να δούμε πώς διάφορες αποφάσεις επηρεάζουν τις αγορές. Στο τέλος, εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε το δοθέ νομικό πλαίσιο. Έτσι θα προχωρήσουμε. Η Μπάνκα Ιτάλια, ίσως αυτό να μου ξέφυγε αυτή η μελέτη, υπάρχει διαφορετικός αντίκτυπος στις τράπεζες από τα MRL. Ένας τομέας είναι οι αγορές, όπου οι τράπεζες και οι χώρες δεν έχουν πραγματική πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίων. Εκεί είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί MRL, εκτός από την κράτηση εσόδων και στεδιακή σώρευση. Μετά, σε αρκετές χώρες Υπάρχουν διαφορετικές τραπεζικές αγορές, υπάρχουν τράπεζες που είναι, χρηματοδοτούνται βασικά από τις καταθέσεις έχουν στοιχεία ενεργητικού, ίσως να μην έχουν ομόλογα, να έχουν καταθέσεις στον ισολογισμό τους. Για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα επίπεδα του MRL, αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Υπάρχουν και διάφορες στρατηγικές εξυγίανσης Ίσως να υπάρχουν τράπεζες όπου η στρατηγική εξυγίανση δεν είναι η πλήρης ανακεφαλοποίηση της τράπεζας, αλλά πώληση επιχείρησης, μεταφορά διαφόρων τομέων. Άρα υπάρχουν διάφοροι τομείς προς εξέταση. Αυτό κάνουμε, ούτως ώστε να είμαστε αναλογικοί. Να πω και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στη ρευστοποίηση σε περίπτωση που αποφασίσουμε ότι δεν είναι εποφελές για το δημόσιο να υπάρξει η διάσωση της τράπεζας, αλλά η εθνική αφαιρεγγιότητα είναι η λύση, τότε το MRL αντιστοιχεί με τις κεφαλουχικές απαιτήσει. Δεν έχει άλλο ένα επίπεδο MRL για αυτές τις τράπεζες. Τέλος, επίπεδο 2 και επίπεδο 3, στοιχεία ενεργητικού επίπεδου 2 και 3 που έχουν περιορισμένη ή δεν έχουν ε, αγορά ρευστού. Αυτά πρέπει να εξεταστούν όπου το SSM παρακολουθεί εκ του ως εποπτικός φορέας και στη δική μας δουλειά το λαμβάνουμε υπόψη εξετάζοντας το σωστό διαχωρισμό, τη δια, ε, τη ρευστοποίηση χαρτοφυλακίων κλπ από την αρχή το έχουμε υπόψη μας αυτό, αλλά είναι κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται από SSM και SRB. Τελευταία παρέμβαση. Take you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μου δώσατε και χρόνο στο τέλος της ε, συνεδρίας. ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σχόλια που έγιναν για την αυξημένη πιθανότητα ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Ως Βρετανοί ούτε και εμείς δεν ξέρουμε το τι θα γίνει, ό,τι ξέρετε ξέρουμε. Αλλά θα ήθελα να αφαιρθώ στο σχόλιο σας για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους, ειδικά στο Λονδίνα, όταν η Κεντρική Τράπεζα πέρσι ε, έκανε προετοιμασίες με κάποια νομικά μέσα όσον αφορά την προτιμησιακή μεταχείριση ε, κρατικών ομολόγων ε, ευρωπαϊκών ε, εν ώψη του Brexit ε, θα μπορούσε αυτό να έχει κάποιες συνέπειες για το εάν και κατά πόσον θεωρούνται τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα μηδενικού κινδύνου. Δεδομένου βεβαίω και του ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι έχουν πολύ μεγάλη έκθεση όσον αφορά την εκαθάριση swap στην Ευρώπη. Δεδομένου του ότι όλα αυτά βρίσκονται υπό το PRA, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα ένα διπλό χτύπημα και για, το κεφα... και για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αλλά και για το πιθανό κούρεμα ε, ομολόγων της Ευρωζώνης ε, όσον αφορά τις κεφαλαιοποιημένες υποχρεώσεις των κεντρικών της Θα ήθελα λοιπόν να μάθω το σχολείο σας για το ότι θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση του Brexit χωρί συμφωνία. Να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, το σχόλιο μου δεν αφορούσε το Brexit, ήταν ένα γενικό σχόλιο ότι δηλαδή η κεντρική αντισυμβαλόμενη είναι στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής μας οπότε θα πρέπει να ξέρουμε το τι θα γίνει. Αυτό ήταν το σχόλιο μου. Για το Brexit χωρίς συμφωνία πρώτα απ' όλα θα έλεγα το εξής. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση συνεργασία ε, με τις Βρετανικές αρχές, ε, δηλαδή στην περίπτωσή μας ε, την Τράπεζα της Αγγλίας. Όπως και με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και έχουμε τώρα τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που θα μας βοηθήσουν στην περίπτωση προβλήματος. Μπορούμε να, μπορούμε να συζητήσουμε και να λέμε το τι θα γίνει σε περίπτωση κουρέματο κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή υποθέτουμε ότι θα βρεθεί ένας τρόπος για να γίνουν τα πράγματα απλούστερα και όχι πιο περίπλοκα. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η πολύ πλούσια ε, ακρόαση. Σας ευχαριστώ κυρία Κένιγκ. για το ότι απαντήσατε πολλές και δύσκολες ερωτήσεις. Βεβαίω, θα πρέπει να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε τον διάλογο μας. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε εδώ με αυτό το θέμα της μερίσιας διάταξης. And we move to the next one. Περνάμε στο επόμενο, Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ και ε, τροπολογίες επί του προϋπολογισμού. Και όπως ε, πάντα, συνάδελφοι, παρακαλώ. We have not concluded our meeting. We have another... Δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Έχουμε ένα ακόμα σημείο και όπως σας έλεγα, πρόκειται και τον προϋπολογισμό που όπως ε, κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζετε επικεντρώνεται κυρίως ε, στον προϋπολογισμό που είναι θέμα που μας αφορά για τα οικονομικά και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Μούρεσαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα συνάδελφοι και να πω και από πλευράς μου επειδή είναι και αρχή της θητείας ε, ότι καλύτερο για την ε, εκπλήρωση των καθηκόντων σας. Ξεκινάμε λοιπόν τον προπολογισμό ε, για το 2020. Όπως γνωρίζετε, ίσως αυτό είναι το τελευταίο έτος για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και στην αρχή του πολιετούς πλαισίου πρέπει να πλαίσουμε τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο για να είναι τελικά έτοιμα να απορροφήσουν τα κονδύλια που τους διαθέτουμε. Και τώρα, στο τελευταίο έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο για να πληρώσουν για τα ποσά τα οποία θα ε, ζητήσουν. Γιατί στην αρχή του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου δεν είναι έτοιμε οι χώρε να απορροφήσουν τα κονδύλια και υπάρχουν καθυστερήσει και στο τέλο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου έχουν αυξήσει τη δυνατότητα απορρόφησης, ε, παρουσιάζουν όρημα προγράμματα υψηλή ποιότητα, αλλά πάντα πρέπει να πληρωθούν και τα χρήματα και τα οποία προέρχονται κυρίω από τη συνεισφορά των κρατών μελών. Η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν τώρα θα είναι να έχουμε μια ένωση η οποία θα μπορεί να εκπληρώσει ε, τις υποχρεώσεις της και να πληρώσει τους λογαριασμούς τους. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο μήνυμα ε, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να πληρώνει τους λογαριασμούς της. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις αυξήσεις που ζητάμε, γι' αυτό και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε ενωμένοι ε, ε, ενώπιον του Συμβουλίου. Ιδίω όταν το Συμβούλιο προτείνει αδικαιολόγητες περικοπές ώστε να μειώσει τα ποσά τα οποία πρέπει να πληρώσουν οι χώρες μέλη στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας δώσω μία μικρή εικόνα του προϋπολογισμού για του χρόνου και όπως έλεγε και ο Πρόεδρος, το τομέα των ενδιαφέροντός μας που είναι κυρίως οι δαπάνες ΕΖΑΣ. Τώρα, το προσχέδιο προπολογισμού που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020 σε απόλυτους όρους σε σχέση με το προσχέδιο προπολογισμού του 2019 έχει αύξηση αλλά σε σχετικούς όρους έχει μείωση σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα της Ένωσης. Πέρσι ήταν 0,00 το ε, καθάριστο χώριο εισοδήματο τώρα είναι 0,99. Σε σχέση λοιπόν με το καθάριστο χώριο εισόδημα έχουμε μείωση, επομένω είναι πάρα πολύ σφιχτό ο προπολογισμό. Παρά το γεγονό ότι είναι σφιχτό, το Συμβούλιο κάνει περαιτέρω περικοπέ. Να σα δώσω κάποια παραδείγματα. Το Συμβούλιο κάνει τις μεγαλύτερες περικοπές στον τίτλο 1α, που είναι ο τίτλος ο οποίος υποτίθεται ότι χρηματοδοτεί την έρευνα, την καινοτομία, τις υποδομές, τομεί δηλαδή οι οποίοι ενισχύουν την οικονομία μας και την κάνουν και πιο ε, ανθεκτική για το μέλλον. Προτείνονται περικοπές 400 εκατομμυρίων ευρώ στον ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομία Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει 200 εκατομμύρια περικοπές στο Connecting Europe Facility, το μεγάλο πρόγραμμα υποδομών, το οποίο πιστεύω ότι χρειαζόμαστε όλοι και μάλιστα προτείνει και 116 εκατομμύρια ευρώ ε, περικοπή στην ε, πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων, που είναι μια πρωτοβουλία την οποία το Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία υπερασπίστηκε ανέκαθεν ε, τα τελευταία χρόνια. εμείς και το Κοινοβούλιο θεωρητικά συμφωνούμε όταν λέμε ότι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία, θέλουμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να επενδύσουμε σε έρευνα, καινοτομία κλπ. Και μετά από τις δηλώσεις, εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε πάντα διατεθειμένοι να αυξήσουμε τα ποσά, όπου βεβαίως είναι δεόντως αιτιολογημένο, διότι όπως είπα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις αυξήσεις, διότι οι δημόσιοι πόροι ε, είναι σε σπάνιδα, αλλά ε, εμείς ε, τηρούμε αυτά τα οποία υποσχόμαστε και να ε, δώσουμε κονδύλια εκεί που χρειάζονται, ενώ το Συμβούλιο προχωράει σε περικοπές και νομίζω ότι αυτό είναι ανησυχητικό. Και γιατί. Διότι όσον αφορά τις ε, τροπολογίες του προπολογισμού, εγώ θα κάνω τις εξής τροπολογίες. Το Συμβούλιο προτείνει μείωση κατά 90 εκατομμύρια ευρώ της ε, εγγύσεις εύση σε σχέση με το προσχέδιο προπολογισμού. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση. Εμπιστεύομαι την ε, ε, εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι χρειάζεται για τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΙ, Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να επανέλθει στο επίπεδο του προσχεδίου προπολογισμού. όχι να το αυξήσουμε, αλλά να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Το ίδιο και με το SRSP για το ε, πρόγραμμα στήριξη. Ε, το οποίο προτείνει το Συμβούλιο να μειωθεί κατά 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι εργαλεία, χρηματοδοτικοί πόροι που βοηθούν τι ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και στήριξη προ χώρε που κάνουν διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. κάτι το οποίο ανέκαθεν υπερασπιζόταν το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν να απορρίψουμε τι περικοπέ του Συμβουλίου για, τις, ε, για το πρόγραμμα στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να επανέλθει στο προσχέδιο προπολογισμού που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο κάνει περικοπέ στον προπολογισμό των ακόλουθων γενικών διευθύνσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τι δραστηριότητε μα. Στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΗΝ, Petition, Ταξούντ, Φίσμα και ΕΣΤΑΤ. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα ποσά τα οποία προτείνουν να περικοπούν είναι τα ίδια ποσά σε επίπεδο όλων των γενικών διευθύνσεων. Αυτό δείχνει σαφώ ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο βασίζεται σε κάποια πολιτική, αλλά είναι ε, ένα συμπέρασμα το οποίο αναζητάει τεκμηρίωση, σαν λογιστική το Συμβούλιο θέλει να απομυζήσει τα πάντα, να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο του προπολογισμού και έχουν πιάσει ένα κόκκινο στυλό και σβήνουν τα ποσά για όλε τι γενικέ διευθύνσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να του επιτρέψουμε να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί για μα ο προπολογισμό δεν είναι καθαρή λογιστική, είναι εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να επιτύχει του στόχου πολιτική τη. Επομένω, αυτέ οι περικοπέ, οι οποίε βασίζονται στι δραστηριότητε αυτών των γενικών διευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν δικαιολογούν και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στο προτινόμενο ποσό του προσχεδίου προπολογισμού της Επιτροπής. Όχι να ψηφίσουν τώρα. Πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Το 2018 εγώ ήμουν γενικός εισηγητής για τον προπολογισμό εξ του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Προπολογισμών. Πρότειμα να γίνει το εξής να υποστηρίξουμε πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις που προτείνουν οι συνάδελφοι που έχουν λάβει Α ή Β από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαθμό. Ξέρετε ότι όλοι έχουμε δικαίωμα να προτείνουμε πιλωτικά προγράμματα προπαρασκευαστικέ δράσει και μετά γίνεται αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Α σημαίνει ότι είναι τέλειο και μπορεί να προχωρήσει χωρί δισταγμό. Το Β σημαίνει ότι είναι καλό και μπορεί να εφαρμοστεί με μικρέ προσαρμογέ. Το Σ και το D σημαίνει ότι το πιλωτικό πρόγραμμα είτε δεν είναι προ εφαρμογή, είτε ήδη καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό προτείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, φέτο να κάνουμε ε, ό,τι κάναμε και τα τελευταία δύο χρόνια, να υποστηρίξουμε δηλαδή τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία λαμβάνουν ε, βαθμό A ή B από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σημαίνει ότι θεωρούνται καλά και μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε και για να σας παραπέμψω και στα ΕΖΑΣ. Εγώ ζητώ κατάλληλη χρηματοδότηση για αυτές τις δαπάνες και φυσικά πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτά τα οποία θέλει ο νομοθέτης. Είναι κάτι ε, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και μετά από διαβούλευση για το μόνιμο, με το μόνιμο εισηγητή για τις ε, εποπτικές αρχές θεωρούμε ότι ο προπολογισμό είναι κατάλληλο. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε, τουλάχιστον αυτό που προτείνεται στο προσχέδιο προπολογισμού και προτείνω να ε, υποστηρίξουμε αυτή τη θέση. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά οι προτεραιότητέ μα είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και υποστήριξη ε, της Νομισματικής και Τραπεζικής Ένωσης και φυσικά να υπάρχει προπολογισμό για την υποστήριξη αυτών των ε, στόχων. Μέχρι τις 25 Ιουλίου, πριν από τις διακοπές, μπορούμε να τροποποιήσουμε τη γνωμοδότηση. Θα ψηφιστεί το Σεπτέμβριο και μετά φυσικά οι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν ε, τροπολογίες επί του προπολογισμού και η Επιτροπή Προπολογισμού ε, τέλος Σεπτεμβρίου θα ψηφίσει όλες τις τροπολογίες. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Όπως θα έκανε και ο πρόεδρος ανέφερε στο χρονοδιάγραμμα, θα τελειώσουμε τις 5, υποστηρίζω πλήρως την αποκατάσταση των προτάσεων του προσχεδίου προπολογισμού. Είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου από τη μία πλευρά να θεσπίζουμε νομοθεσία και να αναθέτουμε στις υπηρεσίες μας και ελληνικές μας διευθύνσεις στόχους και από την άλλη περικόπτουμε τα χρήματα και δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αυτούς τους στόχους. Ελπίζω αυτή η Επιτροπή να είναι ενωμένη και ισχυρή και να ακολουθήσει την πορεία που σκιαγράφησες ανεξάρτητα από τις διάφορες λεπτομέρειες και τις αποκλίνουσες απόψεις θα στη συζήτηση. Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον κύριο Μουρεσάν, τον εισηγητή, για αυτό το σχέδιο κειμένου. Πιστεύω ότι έκανε καλή δουλειά με τα χαρά να ξεκινήσουμε το θεμετικό έργο επεξεργαζόμενο το μελλοντικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το 2020. Λαμβάνουμε αποφάσει όμω ο προπολογισμό είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία μα για να εξασφαλίζουμε ότι εφαρμόζουμε τι πολιτικέ μα. Όπω και στην πρώτερη θητεία, η ομάδα μου επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι δαπάνε για την πρόληψη τη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή αποτελούν ε, επένδυση. Χρειάζονται αυτοί οι πόροι για να υπάρχει η δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτή η δράση θα οδηγήσει σε αύξηση του εισοδήματο για χρηματοδότηση δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, μαζί με του Πρασίνου, Ρηνιού προτείνουν ένα νέο παρατηρητήριο φορολογικό. Ανεξάρτητο παρατηρητήριο με στόχο τη βελτίωση τη πρόσβαση στοιχεία και να κάνει εκτιμήσεις για να δίνει στους διαμορφώνοντες την πολιτική ε, διάφορες, διάφορα στοιχεία και εμπειρίες. Καλούμε τις ομάδες να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία που θα είναι υποφελής για όλους, αλλά πάνω απ' όλα για τους πολίτες ε, της Ένωσης. Επίσης, προτείνω να αυξηθεί η διάθεση των πόρων στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Τον περασμένο Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αυξήσει τις ευθύνες τους και να βελτιωθεί το δίκτυο διακυβέρνησης για την τράπεζα, χρηματοστικές αγορές, τίτλες ασφαλείες, ασφάλειες και συντάξεις. Να βελτιωθεί η λειτουργία του υποπτικού φορέα. Θέλουμε το υποπτικό πλαίσιο να ισχυροποιηθεί στον τομέα της καταπολεμήσεως του ξεπλήματος ε, χρήματος και της χρηματοδοτήσεως των τρομοκρατών. Αυτές οι καλές προθέσεις απαιτούν επαρκείς πόρους. Οι δεμοί θα παραμείνουν απλώς αγαθές προθέσεις. Εν γέννη, ελπίζω οι συγητής και οι υπόλοιποι από τους Σκιώδης να εξασφαλίσουν ότι ο προπολογισμό του 2020 θα λαμβάνει υπόψη τις, τις πρόσφατες απαιτήσει των πολιτών που θα υπάρχουν χρήματα που θα προωθούν δραστηριότητες που θα είναι πιο βιώσιμες και θα καλύπτουν περισσότερους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Λουίς Καρικάνο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον εισηγητή έξοχη δουλειά που έκανε. Συμφωνούμε με την άποψή του. Οι προτεραιότητες ενώσεως και της ομάδας πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους. Ο εξυγχρονισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας η σημασία η καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων, η αλλαγή του κλίματος, όλοι αυτοί οι στόχοι απαιτούν χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει και για τους εποπτικούς φορείς επαρκή χρηματοδότηση και προτείναμε μια υπηρεσία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλήματος του χρήματος και ελπίζουμε ότι και αυτό θα έχει προτεραιότητα στον προπολογισμό. Ένα από τα μέλη μας αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα δοθέντως ότι είμαστε όλοι νέα μέλη. Ο χρονισμός για υποβολή τροπολογιών είναι πολύ σύντομος. Και η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα το Σεπτέμβριο. Μπορούμε να έχουμε κάποια ευελιξία όσον αφορά αυτό το θέμα των τροπολογιών και της ψηφοφορίας ή είναι αδύνατο να αλλάξει κάτι. this Θα το ελέγξουμε. Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Από την πλευρά μας, επίσης, ευχαριστούμε τον εισηγητή για την έκθεσή του. Είναι καλή βάση για τις συζητήσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω τα υποθέτα. Όσον αφορά τον προπολογισμό των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία τη νομοδοτήσεω για να ξεκαθαρίσουμε ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το θέμα. Όταν ο πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Φορέα ανέφερε ότι με τους πόρους που έχει η EBA δεν μπορεί να εκτελέσει του στόχου της για την καταπολέμηση του ξεπλήματο του χρήματο πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Όταν το λέει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τραπεζών. Και βλέποντας και τον προπολογισμό για τις Ευρωπαϊκές Επιτοπτικές Αρχές, θα πρέπει μέσω των ε, γνωμοδοτήσεων να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της χρηματοδοτήσεω. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τις δαπάνες για τη Eurostat. Είναι παλιό το θέμα. Ξέρετε, Πρόεδρε, το συζητήσαμε εκτενώς ε, στα πλαίσια της εκθέσεώς σας. Μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες, από το μεγαλύτερο, ε, τα μεγαλύτερα κονδύλια είναι τα κονδύλια για το Eurostat. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά παρουσιάζουν με φρικτό τρόπο τα στοιχεία. Αν κάποιος απλός άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά που χρηματοδοτούμε, απογοητεύεται θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό για να του πιέσουμε λιγάκι, ούτω ώστε η ιστοσελίδα του επιτέλου να είναι φιλική προ το χρήστη. Ούτω ώστε απλοί φοιτητέ να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία χωρί να χρειάζεται να έχουν πτυχίο στατιστικολόγου. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσει. Παρομοίω, υπάρχει και χρηματοδότηση για την επικοινωνία στον τομέα της Ευρωζώνης. Έχουμε διάφορες ερωτήσεις που μας απευθύνονται, κρίσιμες για τη λειτουργία του ευρώ. Όλοι πρέπει να τα κουβεντιάζουμε αυτά. Με τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα. Κυρίως πιο λεπτομερή επιχειρήματα και πιο φιλικά προς το χρήστη. Στην περασμένη θητεία επεξεργαστήκαμε τους διάφορους λογιστικούς φορείς Είχαμε διάφορα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου πάνω σε αυτό. Είδαμε θετικές εξελίξεις με την ΕΦΡΑΚ. Αλλά δεν είδαμε την ίδια θετική εξέλιξη με το IASB. Υπάρχουν ακόμα κοινοβουλευτικέ απαιτήσει που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συμβολικό ποσό να μπει στο αποθεματικό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε από καλύτερη βάση με αυτού του φορείς και να δεχθούν ε, μια μεγαλύτερη ε, ε, δημοκρατική λογοδοσία. Ευχαριστώ. Γκούναρ Μπέκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σίγητα για τα ξεκάθαρα λόγια σας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, όπως ξέρετε στην ομάδα μας έχουμε μια κάποια ε, διανοητική αντίσταση απέναντι στο αξίωμα του ότι η εναρμόνιση σημαίνει πάντα βελτίωση. Εμείς προτιμούμε να βλέπουμε τον ε, ελεύθερο ανταγωνισμό. Μετά κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις στην παράγραφο 2. Εδώ πέρα γίνεται λόγος για συντονισμό και επίβλεψη των μακροοικονομικών πολιτικών εντός της Ένωσης και των κρατών μελών. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι οι συνθήκες της Ένωσης δεν δίνουν αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν συναρμοδιότητα. Άρα μόνο έναν επικουρικό ρόλο. Οπότε η επίβλεψη μου φαίνεται κάπως να τα ξεπερνάει όλα αυτά. Και τέλος, για την παραγραφό 4. Εκεί πέρα λέτε ότι οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύονται με τα απαραίτητα κονδύλια. Και εδώ να παρατηρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τον ΦΠΑ, τον οποίον διαχειρίζονται όμως τα κράτη-μέλη, ε, δεν έχει καμία δουλειά στα φορολογικά. Σας ευχαριστώ και για την δημιουργική ερμηνεία των ε, συνθήκων, αλλά σας διαβεβαιώ πως η πολυμερής εποπτεία είναι το άρθρο 121 και 126. στο άρθρο 5 επίσης ε, ε, η οικονομική πολιτική δεν είναι επικουρική αρμοδιότητα, είναι μια αρμοδιότητα συντονισμού και πολλοί αρμόδιοι θεωρούν ότι είναι συναρμοδιότητα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που δεν θα κάνουμε σήμερα όμως. Ντέρκ Γιάν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Με χαρά μου λέω ότι μπορώ και εγώ να στηρίξω την έμφαση που αποδίδει στις ποιοτικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Όμως Βεβαίω, όπω πάντα, ο διάβολο κρύβεται σε λεπτομέρειε. Το ECR είναι υπέρ ε, τη δημοσιονομική μετριοπάθεια. Θα θέλαμε να υπάρξει εξορθολογισμό. Η λογοδοσία επίση έχει μεγάλη σημασία για να έχουμε αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και πραγματική αξία. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, πράγματι ε, στην αναθεώρηση υπάρχει ε, μια στελέχωση. Δεδομένου του ότι η τελική συμφωνία επετεύχθη πολύ βιαστικά θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε προσεκτικά το τι σημαίνουν αυτά. Θα πρέπει να συνεχίσουν να λογοδοτούν οι ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ. Τέλο, κύριε Πρόεδρε, με χαρά βλέπω πω ο εισηγητή συμπεριέλαβε την πρόταση του Συμβουλίου για την ε, πρόσθεση ενός λεπτομερούς παραρτήματος από την Κομισιόν που θα αυξήσει κατά πολύ την διαφάνεια και την λογοδοσία. Ευχαριστώ εσάς και τον εισηγητή λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριος Γκουσμάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνούμε με την άποψή του. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί με τις περικοπές που προγραμματίζονται εδώ. Πρέπει να ανησυχούμε και να δούμε τις ε, επενδύσεις. Οι περικοπές ε, στην έρευνα, στην καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, πάνε σε λάθος κατεύθυνση και στην αντίθετη κατεύθυνση από τις συστάσεις της Κομισιόν. Και όταν μιλάμε για λεφτά τα οποία επενδύονται στην καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, είναι επενδύσεις. Είναι λεφτά τα οποία θα αποδώσουν. Και το ίδιο ισχύει και για την κλιματική αλλαγή. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να περιέχεται σε όλα τα έγγραφα διαμόρφωσης πολιτικής ε, και της πολιτικής του προπολογισμού και βεβαίως ε, τα ζητήματα μακροοικονομικών ανισορροπιών και της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σίγητης ε, θέλει να απαντήσει. Γρήγορα παρακαλώ. Όχι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να σας πω ότι αναμένω την συνεργασία μας ε, με τρόπο που θα κατανείμει σωστά τους πόρους, να ενισχύσουμε την οικονομία, την απασχόληση στην Ευρώπη και να έχουν και εποπτικές αρχές ε, αρμοδιότητός μας όλους τους πόρους που χρειάζονται και να βρούμε βέβαια τη σωστή ισορροπία ε, μεταξύ της επάρκειας πόρων ε, και της επίτευξης των στόχων που έχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για το χρονοδιάγραμμα. Δύσκολα φαίνονται τα πράγματα για την επέκταση της προθεσμίας. Μπορούμε να την αναβάλουμε μέχρι τις 5 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι. Να κερδίσουμε 5 ώρες. Μου λένε ότι αυτό είναι το καλύτερο που γίνεται. Οπότε, η προθεσμία είναι 25 Ιουλίου, 5 το απόγευμα, για τροπολογίες ε, και ε, για τις γραμμές του προπολογισμού. 4 Σεπτεμβρίου θα εξεταστούν αυτές. Ορίστε. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος της Επιτροπής Ήτρε, εγώ ξέρω πως η προθεσμία είναι 5 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται αυτό εδώ. Α, γιατί εμεί πρέπει να ψηφίσουμε στις 4 Σεπτεμβρίου, λέει ο πρόεδρος. Έτσι, τότε ψηφίζουμε. Οπότε με την ψηφοφορία πάει. Τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Επόμενη συνεδρίαση, όπως ξέρετε, είναι ακριβώς στις 4 Σεπτεμβρίου και 5 στις 4 είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε ακρόαση της υποψηφίου για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της κυρίας Λαγκάρντ και άλλα πολύ σημαντικά θέματα και τον προπολογισμό βεβαίω. Αρκετά σημαντικός και αυτός. Και ψηφοφορίες λοιπόν. Ακροάσεις, Ενρία, Λαγκάρντ, μέρτ και αργά το απόγευμα ψηφοφορίες για τις θέσεις της ΕΚΤ και για τον προϋπολογισμό. Λύεται λοιπόν αυτή η συνεδρίαση. Καλές διακοπές. Μετά την προεκλογική εκστρατεία χρειάζεται και λίγη ξεκούραση ε, για να χαλαρώσουμε και να επανέλθουμε δυναμική ε, από Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελίτη συνεδρίαση.